Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ καθίστε και προετοιμάστε τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας. Έχουμε πολύ συναρπαστικά θέματα για να ψηφίσουμε σήμερα. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά και να συμφωνήσουμε σε όλα. Οπότε... Λοιπόν, θα τα λέω σιγά για να βρείτε όλοι τις κάρτες σας, ετοιμαστείτε, γιατί είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οπότε, ψηφίζουμε για την προφορική ερώτηση για την κλειφωσάτη. Μία ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Το ελπίζω. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Στο επόμενο πάμε. Γρήγορα. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση. Έχει αρκετέ ε, τροπολογίες. Πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέταρτη τροπολογία υπέρ, κατά, Εμένα μου φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά να το ξαναδούμε. Τροπολογία 4. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 5 καταπίπτει, τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία και πέρας και εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την εντολή ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Τώρα ψηφίζουμε για την έκθεση για τον καταμερισμό των προσπαθειών συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές πριν ψηφίζουν οι σοσιαλιστές, συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. δώδεκα και άγκρι δεκατρία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 17 υπέρ. Κατά. Να το Η Ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία και πέρας. απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να την επολιτεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Πού πάμε. Συμβιβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Τροπολογία 142. 142 υπέρ. Στη λίστα μου έχουν δώσει εδώ τη γραμματεία ψηφίζουμε την 142. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141. Και 65. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πού πάμε. Ε, γυρίστε μερικές σελίδες. Εκεί. Πολλές σελίδα 20, τροπολογία 194. Σε δικιά μου τη λίστα είναι σελίδα 20. Λοιπόν, 194 υπέρ. Δεν τη βρήκατε. Περιμένω λοιπόν. 194. βρήκατε. Ποιο ποιος είναι ο Σκιώδης στο ΕΛΚ. 1-9-4. βρήκατε. Κυρία Αγιούζο, άμα τη βρείτε πείτε μας. Σελίδα 18 στη λίστα του ΕΛΚ. Ε, δεν καταπίπτει μου λένε εδώ. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ήταν στην εναλλακτική συμβιβαστική που δεν εγκρίστηκε. 194. Το βρήκε η κυρία Γιούζο. Λοιπόν, υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Ναι, κατά. Απορρίπτεται. Πάλι γυρνάμε μερικές σελίδες. Τα έχετε καλύψει όλα. Τη συμβιβαστική. Συμβιβαστική C. Σελίδα 30 μου λένε εδώ. Υπέρ τη συμβαστική C. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.46 και 29. να έχει γίνει αυτό. Μάλιστα. Να, εντάξει. 25 και 26 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.48 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 30 και 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνονται. 2.50. 2.55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Όχι. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε μερικές σελίδες. Ήτρε 35. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. άλλη μια σελίδα πιο εκεί, ήτρε 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεν έχω δει το ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ, ευχαριστώ, κατά, αποχές, να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. Εγκρίνεται. Ήτρε 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά Εποχές εκκρίνεται. Μάλιστα. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται μάλιστα. 44 καταπίπτει 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τοπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τραν καταπίπτει. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται. Έξι της Επιτροπής Μεταφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη γυρνάμε πάλι μερικές σελίδες, τροπολογία 10, πολλές σελίδες. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ της 99. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να την επαληθεύσουμε. Τραν 8. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά εποχέ απορρίπτεται. Και μετά έχουμε την τελική ψηφοφορία το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κύριε Γκερμπράντι, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχουμε τώρα μία δύσκολη απόφαση αν θα ζητήσουμε ψήφο, για ψηφοφορία για εντολή. Δεδομένων των συνθήκων αποφάσισα να μην ζητήσω κάτι τέτοιο, τέτοια ψηφοφορία. Ε, δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να πάμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. next vote... Επόμενη ψηφοφορία για τη σήμανση στη διάθεση προϊόντων λίπανσης και την τροποποίηση του κανονισμού της Επιτροπής. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκαρντίνη. Ψηφίζουμε. Είστε έτοιμοι. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207-211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 209 και 210 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Να την επαληθεύσουμε γιατί 209 και 210 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6. Τροπολογία 6. Περ. Κατά. Επαλήθευση. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 217. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Και πάλι υπέρ της 9. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221-222 υπέρ. Κατά να την επαληθεύσουμε. 221-222. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνονται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές οι φιλελεύθεροι δεν σηκώνουν το χέρι τους πρέπει να παρηθεύσω λοιπόν τη 227 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση για την συμβαστική τροπολογία 15. Πέραση της Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ Α, συγγνώμη, 235 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε τη 236. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 237, 238, 39. Ποιος είναι υπέρ αυτού του μπλοκ τροπολογιών κατά αποχές επαλήθευση για τον μπλοκ. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτονται. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ναι, πέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. 244. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 250. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 252. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 254 επαλήθευση. Επαλήθευση της 254, πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 255 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε μερικές σελίδες. 291. Υπέρ της 291. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε, γιατί το ECR δεν είδε να σκόνει τα χέρια του. 2,91. Ήσασταν κατά, πέρα της ψηφοφορίες, απορρίπτεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 292. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 και 293 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 294 καταπίπτει. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 317-318. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 320. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 321-322 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 334 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 335 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 336 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση. Για την 336. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Για την 16. Πέραση της ψηφοφορίες, Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. τις 17. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 345. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 350-351 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, συγγνώμη, 22 υπέρ, υπέρ της 22, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Της 26. Πέραση της ψηφοφορίας. Συγγνώμη, περιμένω. Επαλήθευση της 26. It's okay. Everyone voted, so... Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 362 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. 365, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία με την προηγούμενη. 367 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 368-369 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 370 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 371 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 372 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 και 373. Α, αυτές οι δύο καταπίπτουν γιατί εγκρίναμε μια τροπολογία κάποια στιγμή. 374. Υπέρ. Της 374. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά να το επαληθεύσουμε. Για την 374. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 32 και 375. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε ε, αρκετές σελίδες παρακάτω στην 430. Υπέρ της 430. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. 430. Σχεδόν Τελειώσαμε. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 429. Περ. Τη 429. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 431. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 432. 433. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 435, 400, συγγνώμη, 434 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 435, 436, α, συγγνώμη, ήταν όλες μαζί. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 443 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για τη 41. Αλλάζετε γνώμη συνεχώς και αλλάζει το μπλοκ πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 444 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 451-452 υπέρ, κατά, αποχές, 451-452 να επαληθεύσουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 455 υπέρ. 455 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 445 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές 42 πάλι υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές απορρίπτεται. 43-446 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44-447 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 45-448 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 449 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 450 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 450. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 463 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 465 υπέρ κατά, αποχές, επαλήθευση. Δεν σηκώσατε τα χέρια σας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 464 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 466 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 510 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 511 υπέρ. Θέλετε επαλήθευση για την 510. Να επαληθεύσουμε. The vote is και απορρίπτεται. 511 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 513-514 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 512 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 515 υπέρ, κατά, Ας την επαληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 515, 516 υπέρ. Με συγχωρείτε, 517 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 518 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 519 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 520 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 521 και 522 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 523-524 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 525 και 526 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 527 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 528 απορρίπτεται. 529 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 και 530 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας την ελέγξουμε. 50 και 530 επαληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 531-532. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 533 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ήταν σαφές. Και ψηφίζουμε ξανά 533-534 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 51 και 535 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 και 536 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 537-538 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 53 και 539 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 και 540 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 541 υπέρ κατά απορρίπτεται 56 και 542 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 543-544 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 545 υπέρ κατά απορρίπτεται 546 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 547 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 548-549 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 550-551 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 552 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 553 απορρίπτεται 555 και 556 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 554 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 558-557 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57, 559 και 560 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 561 και 562 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59, 563, 564 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 565, 566 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 και 567 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 και 568 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 και 569 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 και 570 απορρίπτεται 571 υπέρ κατά εγκρίνεται για να επαληθεύσουμε στην 571. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 572. Υπέρ. Εκπίπτει. 574 υπέρ κατά απορρίπτεται 575 576 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 577 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 578 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11b υπέρ

κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 593 υπέρ κατά 593. Απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 596 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 597 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 598 599 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 600 εγκρίνεται 603 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 604 υπέρ κατά και αποχές απορρίπτεται 605-606 εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 και 73. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 612 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 613 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 614 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 615 απορρίπτεται. 616 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 617 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 απορρίπτεται 618 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 619 μέχρι 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 623 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από το 624 στο 627 απορρίπτεται 628 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 635 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 637 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 636 υπέρ κατά εγκρίνεται. 638 υπέρ κατά. Θα την επαληθεύσουμε την 638. Πέρας ψηφοφορίες εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. μπλοκ από 639. Το βλέπετε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 646 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 647 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 648 υπέρ κατά απορρίπτεται. 649, 650 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 649-650. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο άλλο έχουμε έναν περισσότερο. Πέρας ψηφοφορίες και εγκρίνεται. 651 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 652 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 653 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 654 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 655 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 656 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 Απορρίπτεται. 660. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία σε μπλοκ από την 661 στην 664. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 665. Υπέρ, κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 675 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 676, 677 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. blog από το 678 ως το 681 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 682-683 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 684 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είμαστε στην 97. Απορρίπτεται. 685 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 686 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπλοκ από τα 687 ως τα 691 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 692 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 693 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 694 Εγκρίνεται. 695 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 696 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 697 Απορρίπτεται μπλοκ το 698 ως το 702 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν μιλάτε. Εκατό. Πάμε λοιπόν στο 100. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 703-704. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 505 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 706 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 707 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 708 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101. 709 και 710 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 713 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 714 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 515 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 716-717 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 719, 720, 721 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Την επαληθεύουμε την 103 What did I say? It's adopted. εγκρινεται Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 722-723 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 724 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 725 υπέρ κατά «525 ξανά πάμε. Υπέρ κατά Άρχεται η ψηφορία την 725. Πέρας. Και απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 726 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105, 727 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106, 728, 729 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 107 δεν την ψηφίζουμε με συγχωρείτε 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 730 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 731 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας την ε, επαληθεύσουμε την 110. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 732 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προχωράμε μερικές σελίδες. Πάμε στην 765. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 766. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...768, 769 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 770 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 771 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 απορρίπτεται 772 υπέρ κατά Ας επαναλάβουμε 772 ποιοι είναι υπέρ εγκρίνεται 773 υπέρ κατά θα ελέγξουμε επαλήθευση 773 πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται 774 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 775 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 776 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 777 και 778 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 779 Απορρίπτεται. 780 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και απορρίπτεται. 781 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 784 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 785-786 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 787 υπέρ κατά κατά απορρίπτεται 788 υπέρ κατά Απόρριπτεται. 789 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 790 791 απορρίπτεται. απορρίπτεται. 791 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 794 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 795 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 796 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 796 797 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 798 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 799 800 και 801 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 802 και 806 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 802-806 υπαλληθεύουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 805. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Το ECR τι κάνει, λοιπόν, 132 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 807 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35-808 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 809 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137-810 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 810 υπέρ κατά απορρίπτεται 812 απορρίπτεται 813 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 814 απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 815 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 816 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 απορρίπτεται. 817 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 818 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 819 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 820 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 821 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 822 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 823 825-824 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 826-827 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 829-830 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας το επαναλάβουμε. 829-830. Ναι, εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131. 832. Απορρίπτεται. 833, 834, 835 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 836, 837, 838 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 839 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 840 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 841 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 842 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 844 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 845 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 846 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 847 και 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 849 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 850 δεν το ψηφίζουμε 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 146 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 147 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 148 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε. στην 161 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181-82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πρέπει να μου το πείτε από την αρχή να τα απορρίψουμε όλα. Οπότε η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας και εγκρίνεται. Α, δεν τελειώσαμε. Μάλιστα. Τώρα ψηφίζουμε HIV, AIDS, ε, φυματίωση και υπατήτηδα γάμα. πατήτε C. Έτοιμοι. Ναι, είναι σύντομο αυτό. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38, 39 42, 43, 44 το σύνολο όχι μόνο αυτά τα δύο 38-39 λοιπόν κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα περνάμε στις 42, 43, 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται.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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την 85 πήγαινε αυτή 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87, 89 και 88 όχι, όχι 87 και 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 καταπίπτει ωραία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές ε, κατά, ε, απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 20 και 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 17 έχετε αντίρρηση για να ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία όχι λοιπόν έχουμε την 17 όπως τροποποιήθηκε υπέρ Κάτι λέει η Τζίνα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22-23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα διορθωθεί αμέσω. Και αναρωτιόμουν, είναι μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και εγκρίνεται. Ωραία. Αυτά αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Τελειώνει εδώ η ψηφοφορία. Okay, business. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η εξέταση ενός σχεδίου έκθεσης. Η κυρία Γκέρλινγκ είναι η συγγήτρια για τη συνέχιση των περιορισμών του πεδίου εφαρμογή για τις αεροπορικές δραστηριότητες. Να δώσω αμέσως το λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια την κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι στην Επιτροπή γνωρίζουν το ιστορικό, δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα-δυο πραγματάκια. Το 1,3 των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από τις διεθνείς αερομεταφορές. Με την αναμενόμενη αύξηση τη και κυκλοφορία κατά τι επόμενε τρει δεκαετίε, οι παγκόσμιε εκπομπέ θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω κατά 300 με 700% έω το 2050, εάν τεληφθούν μέτρα για να συγκρατηθεί η αύξηση. Η ανάπτυξη ενό παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου ω μέρο μια δέσμης μέτρων που προορίζεται να αμβλύνει τι επιπτώσει των εκπομπών από αεροσκάφη επί τη κλιματική αλλαγή, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο θεματολόγιο του Διεθνού Οργανισμού Πολιτική αεροπορία εδώ και κάποια χρόνια. Κατά την 37η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης ε, το 2010, ε, συμφωνήθηκε ένας παγκόσμιος φιλόδοξος στόχος της ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2020. Τρία χρόνια αργότερα ο οργανισμός συνέστησε ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη και την επίτευξη αυτού του στόχου στις 6 Οκτωβρίου του 2016, κατά τα 31 η Σύνοδο, ο ΔΟΠ ενέκρινε την απόφαση 39 39-3, η οποία εισάγει ένα παγκόσμιο σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης ανθρακούχων εκπομπών για τις διεθνείς αερομεταφορές, το Κορσία. Στο πλαίσιο αυτού, οι φορεί εκμετάλλευση αεροσκαφών που σημειώνουν υπέρβαση των εκπομπών θα πρέπει να αγοράζουν αντιστασμιστικέ μονάδε ώστε να το θετερότητα ω προ τι ανθρακούχε εκπομπέ από τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία από το 2021. Αυτή η γραμμή βάση θα υπολογιστεί ο μέσο όρο των εκπομπών τη περίοδου 2019-2020. Το σύστημα έχει σκοπό να συμπληρώσει νέε τεχνολογίε, λειτουργικέ βελτιώσει και μέτρα υποδομή με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη για τι αεροπορικέ μεταφορέ καθώς και το φιλόδοξο μακροπρόθεσμο στόχο του κλάδου για μείωση κατά το ίμιση των καθαρών εκπομπών μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσχωρήσουν στο σύστημα από την αρχή. Ο ΔΕΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα εργαλεία εφαρμογή τα οποία θα επιτρέψουν στο Κορσία να τεθεί σε ισχύ το 2021, τα οποία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα κριτήρια αντιστάθμιση και επιλεξιμότητας, τη εκπομπής γραμμή βάση, καθώ και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συμμετέχοντα κράτη για την υλοποίηση του συστήματο σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια το σύστημα θα υλοποιηθεί σε τρεις ε, στάδια. Κατά τη διάρκεια του πιλωτικού σταδίου 2021-2023 και στο πρώτο στάδιο 2024-2026 θα συμμετάσχουν 65 χώρες σε θελοντική βάση. Στο δεύτερο στάδιο, 2027-2035, με εξαίρεση χώρες με ελάχιστε αεροπορικές δραστηριότητες, θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή. Σε περίπτωση που το σύστημα επιτύχει τους στόχους του, περίπου το 80% των εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών άνω των επιπέδων του 2020 θα αντισταθμίζεται βάσει του Κορσία μεταξύ του 2021 και του 2035. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συμφωνία προβλέπει επανεξέταση κάθε τρία χρόνια, ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος και τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό τον αντίκτυπο των εκπομπών των αεροσκαφών στην αλλαγή του κλίματο και για να δοθούν κίνητρα σε αεροπορικέ εταιρείε να έχουν αποτελεσματικότερου στόλου, εγκρίθηκε νομοθεσία το 2008 για την επέκταση του συστήματο εμπορία εκπομπών στι εκπομπέ σε πτήσει προ, από και εντό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτή η προσέγγιση κρίθηκε συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κάποιες τρίτες χώρες και αεροπορικέ εταιρείες αντιτάχθηκαν στεναρά στην νομοθεσία υποστηρίζοντας ότι ένα περιφερειακό καθεστώς θα οδηγούσε σε αποδυναμωμένες εμπορικές και οικονομικές τρευλώξεις. Στρεβλώσεις. Για να υποστηρίξουμε λοιπόν τη δέσμευση του ΔΟΠΑ για την ανάπτυξη ενό παγκόσμιου και μέτρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να προερορίσει προσωρινά το πεδίο εφαρμογή ε, εντό του ΕΟΧ μέχρι το 2016. Ελήψη περαιτέρω τροποποίηση οδηγία ε, η παρούσα παρέκκληση θα πάψει να ισχύει και θα, ε, επανέλθει η αρχική κάλυψη συμμόρφωση του 2008 γνωστή σε όλου ω snapback. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη Συμφωνία Κορσία το Φεβρουάριο του 2017 και πρότεινε τη διατήρηση της παρέκκλησης πέραν και του 2016. Η περαιτέρω επανεξέταση του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών θα γίνει σε συνδυασμό με την έκθεση της Επιτροπής, ε, δεν προσδιορίζεται πότε ε, και δεν ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη σεφαιώνη από τη ΔΟΠΑ σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο των απαραίτητων μηχανισμών για την εφαρμογή του Κορσία και θα μπορούμε να προσδιορίσουμε το ακριβές περιεχόμενο της συμμετοχής των τρίτων χωρών. Η πρόταση τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ταχεία συμφωνία μεταξύ των δύο συνομοθετών, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2017, ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και συμμόρφωση στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Τώρα, τι κάνει το δικό μου σχέδιο έκθεσης και ποια είναι η διαφορά με το πρόταση της Επιτροπής. Να πω ότι εγώ συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την προσέγγιση θεωρώ ότι σωστά θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο Κορσία να υλοποιήσει τους στόχους του, αλλά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ε, είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση και αυτό κατά την άποψή μου αντανακλά και η έκθεσή μου. Καταρχάς να υπάρχει συνέπεια λοιπόν με την κείμενη νομοθεσία Θεωρώ ότι η παρέκκληση αυτή θα πρέπει να είναι περιορισμένη και σίγουρα θα πρέπει να εκπνεύσει πριν ε, την έναρξη λειτουργία του Κορσία τον Ιανουάριο του 2021. Δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ημερομηνία δημοσίευση 1η ε, Ιανουαρίου του 2019 για την ε, έκθεση εφαρμογή επιτροπή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για το θέμα αυτό και τρίτον πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει εγκαίρως προτάσεις ως απάντηση στην έκθεση εφαρμογής. Επομένως χρειαζόμαστε ημερομηνία για την υποβολή της έκθεσης και, υποβολή για, ε, και ημερομηνία για τις επόμενες προτάσεις. Τώρα, για την ίδια την έκθεση θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για μελλοντική νομοθεσία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα βασικά τεχνικά στοιχεία. Δεν μπορούμε αυτά να τα έχουμε ασαφώς. Η έκθεση θα πρέπει να εξετάσει τη συνολική φιλοδοξία του Κορσία σε σχέση με τι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύστημα εμπορία εκπομπών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα επανέλθω τόσο λίγο. Διότι ε, κατά την άποψή μου αυτό είναι θέμα αρχή. Δεν θα πρέπει να βρεθούμε σε θέση ε, κατά την οποία θα αποδημώσουμε την παρούσα θέση μας. Ε, θα Πρέπει λοιπόν ε, για να συνεχιστεί το σύστημα εμπορίας εκπομπής ως έχει, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ό,τι προτείνουμε θα έχει τουλάχιστον ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή και περισσότερα αν γίνεται. Για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική η έκθεση θα πρέπει να καθορίζει και το επίπεδο συμμετοχής των τρίτων χωρών, τη μεθοδολογία για τη συμμόρφωση, για τις καιρός για τη συμμόρφωση, για τη μη συμμόρφωση, διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, πρότυπα παρακολούθησης, ε, διαφάνεια, ε, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση και κανόνες σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ε, σημεία, η έκθεση εφαρμογή θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στου νομοθέτε να εξασφαλίσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα του συστήματο εμπορία εκπομπών. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα της διαφάνειας και ξέρω ότι πολλά μέλη που συμμετείχαν μαζί μου στην Επιτροπή και στις αποστολές ε, στη ΔΟΠΑ πέρσι, ε, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα ε, για την πρόσβαση σε πληροφορίες από τη ΔΟΠΑ, κυρίως ε, για το CAEP, που είναι η Τεχνική Επιτροπή Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, και εκεί υπήρχαν συμφωνίες μη δημοσιοποίησης των στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι παρατηρητής, δεν έχει από τεχνική σκοπιά δικαίωμα να γνωρίζει καθόλου τι συμβαίνει σε αυτές τις συνεδριάσεις, γιατί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν έχουν υπογράψει ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν πληροφορίες. Και αυτό φυσικά δυσχεραίνει τα πράγματα, γιατί εκεί ε, επελέγει η ε, ανάπτυξη του Κορσία και επομένως εμείς είμαστε σε δύσκολη θέση. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το αναφέρει η έκθεση και προσπάθησα να το αναφέρω μέσω κάποιων τροπολογιών μου. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια Και θα ήθελα να σταθώ και στη δυνατότητα του Κορσία να υλοποιήσει τους στόχους ε, αποταμίευσης και μη χρήσης άνθρακα που θέλουμε. Καταρχά, θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση των καυσίμων. Το Κορσία χρησιμοποιεί μια πιο, ευέλικτη μέθοδο μέτρησης του καυσίμου ε, σε σχέση με αυτή που επιτρέπεται από το σύστημα ETS. Ε υπάρχει ε, αυτή η έννοια της ώρας αναπλόκ, ε, που είναι ένα μοντέλο που μετρά το καύσιμο ανά ώρα, ενώ εμείς στο ETA ε, ζητάμε ε, στοιχεία για το ακριβές καύσιμο που καταναλώθηκε. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι εφικτό βέβαια να έχουμε το ακριβές καύσιμο που καταναλώθηκε. Αυτά βέβαια θα πρέπει να τα δούμε ακόμα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί το θέμα αυτό εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και επομένω και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ε, όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, ε, το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, απαιτεί παρακολούθηση των εναλλακτικών καυσίμων και αυτό ε, την χάνει διαχείριση σε επίπεδο αεροδρομίου. Αυτή τη στιγμή το Κορσία δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο. Επειδή όμως ε, τα εναλλακτικά καύσιμα είναι πολύ σημαντικό θέμα και το έχουν τονίσει στο ε, σύνολο των μέτρων που προβάλλουν στο ΔΟΠΑ, θα πρέπει να ζητήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης. Όσον αφορά το Μητρό, το σύστημα ε, της εμπορίας εκπομπών έχει ένα δημόσια προσβάσιμο μητρό δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην ε, πρόταση του Κορσία και πάλι λοιπόν ε, προβλέπω ότι θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και στο σημείο αυτό και υπάρχει φυσικά και το σαφές νομικό θέμα ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι πολύ εύκολο, βασίζεται στο κείμενο ευρωπαϊκό δίκαιο, το Κορσία βασίζεται σε κάποια διεθνή σύμφαση και επομένως ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι διαφορές που υπάρχουν ε, θα πρέπει κάπως να επιληθούν και να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ε, ε επιμένω αλλά, σε αυτά τα σημεία, αλλά είναι βασικά σημεία διαφοράς αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το σύστημα και θα συζητηθούν σε μια τεχνική συνεδρίαση του ΙΣΤΟΠΑ στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Η ιδέα είναι ότι θα υπάρχει ένα σχέδιο κειμένου έτοιμο για να στείλουν στο Συμβούλιο ε, το Σεπτέμβριο και αυτό στη συνέχεια ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί. Ε, μέχρι λοιπόν το φθινόπωρο φέτος θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς ε, θα κάνει ο ΔΟΠΑ και τι θα προτείνει για τα θέματα αυτά Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια για την έκθεση αυτή αντίστοιχα κάπου τότε κι εμείς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί, αλλά ελπίζω τα μέλη να συμφωνήσουν μαζί μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, μια εύρωστη παράλληλη πορεία με τη διαδικασία του ΔΟΠΑ. Ε, θα μπορούσα να πω βεβαίως πολύ περισσότερα, δεν θα τα πω. Και θα σταματήσω εδώ και προσβλέπω στα όσα έχουν να πούνε οι συνάδελφοι. Uh, Λόγω στον κύριο Λίζα, σκιώδη ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέρλινγκ ε, για το σχέδιο έκθεση. Η είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Ε, είναι κάτι πολύ ευχάριστο να ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς Οι εκπομπέ, ε, διοξιδίου του Αφρικα είναι πολύ ψηλέ από τα αεροπλάνα. Αν υπολογίσουμε τα 129 κράτη, τα οποία ε, επικέψαν τη συνθήκη του Παρισίου, Αυτά τα 129 κράτη παράγουν τεράστιες εκπομπές υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία, η Φιλανδία, ε, η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία και η Σουηδία. Και αν λέγαμε ότι αυτές οι χώρες, Σουηδία, Ουγγαρία, Φιλανδία κτλ. Και άλλες 124 χώρες δεν έχουν συνολικά μαζί τόσες πολλές εκπομπές. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις και αξιώσεις όπως έχουν άλλες χώρες. 129 χώρες και αυτές οι βιομηχανικές χώρες που ανέφερα παράγουν τόσα ε, επικίνδυνα αέρια και γι' αυτό έχουμε μια αποστολή τον Οκτώβριο προηγούμενου έτου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε και ανέκρινε το κόρζι, αλλά εκφράζοντας μια απογοήτευση παράλληλα, το οποίο θα πρέπει να το πούμε με σαφήνεια και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ακόμα ένας διάλογος να μην ε, επαναρθούμε στο παλιό σύστημα εμπόρια ε, εκπομπών. Και μπορώ να πω ότι ε, το πεδίο εφαρμογής είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί αφορά και τον ε, τομέα του ανταγωνισμού. Αν δεν εγκρίνουμε κάποια πρόταση, τότε έτσι θα παραμείνει ότι θεωρώ ότι είναι μια πολιτική αστοχία. Ξεκινήθηκε και γίνανε κάποιες πρόοδοι, πρέπει να τις λάβουμε υπόψη αυτές και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω πάρα πολύ το, την πρόταση της ε, κυρίας Γκέρλινγκ γιατί καθορίζεται μέχρι το 2020 θα πρέπει να παρατείνουμε τη διαδικασία και ότι δεν θα πρέπει να το παρατείνουμε χωρίς κάποια όρεση, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση μέχρι το 2020 και μετά να συνεχίσουμε. Θα ήθελα πιο ε, ακριβή διατύπωση ως προς τις προσδοκίες μας και από ποιους όρους είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε παράτηση και μετά το 2020. Τι μπορεί να μας προσφέρει το Κορσία για να έχουμε μια συνέχεια στις ε, χώρες εντός ε, της ε, Υπηρού. Ποιος θα συμμετάσχει σε αυτό. Μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις ΗΠΑ. και όταν σε κάτι συμμετέχουν το 90% των χωρών ε, της γης, για ποιο λόγο να μην συμπεριληφθεί και να συμπεριληφθούν και οι ΗΠΑ, θα μπορούσε να πει κανεί. Όσον αφορά τα offset του συμψηφισμού, είναι ένα κουτί Πανδόρα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα συμβεί με αυτό, τι, τι σημαίνει αυτό για τη βιομηχανία, να είμαστε σαφείς ότι θα προσδώσει ποιότητα στον κλάδο. Άρα χρειάζεται να το παίρνει μια πιο ε, την τύπωση για τον, ε, την προθεσμία του 2020 και τι θα ισχύσει στη συνέχεια για τις ε, τις τη εντός της Υπήρου. Όσον αφορά το σύστημα εμπορία εκπομπών, θα πρέπει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μια διάρκεια σε αυτό με μεγάλη ε, πλειοψηφία συμφώνησε το Ευρωκοινοβούλιο ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και ε, να συμπεριληφθούν και οι πτήσεις με το 2021 από την Επιτροπή για τις Συγκοινωνίες με τον συντονιστή από το ΕΛΚ ε, έλαβα ένα ακόμα πολύ σημαντικό επιχείρημα συγκεκριμένα ότι ο ανταγωνισμό είναι πολύ ψηλό τη Ευρώπη και ότι δεν αγγίζει πολύ ιδιαίτερα το σύστημα αυτό, των κλάδων τη αεροπορία. Στο πνεύμα βέβαια το περιβαλλοντικό πάντο και γι' αυτό θα ήθελα να ελέγξω τι θα γίνει στο μέλλον και αν θα ε, δραστηριοποιηθεί και το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Άλλη μια πρόταση που θα ήθελα να ε, επεξηγηθεί ε, στο ΕΛΚ και που θέλω να υποστηρίξω. Αν επιβαρύνουμε τις πτήσεις στην Ευρώπη, τότε θα μπορούσαμε άλλες μηχανίες, όπως είναι η χαλιβουργία και τα λοιπά, όπου πρέπει να βοηθήσουμε με απαραίτητους, όπου δεν υπάρχει carbon leakage, διαρροή άνθρακα, αυτό το θέμα το επεξεργαστήκαμε επιστημονικά. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που μπορούν ε, να σας τα επεξηγήσουν, αλλά θέλω να ε, επαναφέρω την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας σωστός, ισότιμος, λογικός καταμορισμός ανάμεσα στην βιομηχανία και στις αεροπορικές πτήσεις. Αν θέλουμε να καταργήσουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών, τότε δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. κανείς δεν μπορεί να έχει αυτή την απέτηση ότι ως Ευρωπαϊκή πρέπει να αποδεχτούμε κάτι που δεν συμφωνηθήκε στο Παρίσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Ντάνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την συγγήτρια και τον κύριο Λίζα για τα σχολεία της. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα θα είμαι πιο σαφής για τις επιφυλάξεις της ομάδας μας για τα μέτρα της ε, Κόρσια. Ε, μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος ε, αποτελεί μεγάλο ποσοστό των εκπομπών και με τις τωρινές προβολές υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστούν οι εκπομπές από το, τα επίπεδα του 2010 μέχρι το 2050 και βεβαίως έτσι υπάρχει ο κίνδυνος ε, υπονόμευσης όχι μόνο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά των παγκοσμίων προσπαθειών για τις δεσμεύσεις ε, του Παρισιού. Βεβαίως ε, η φιλοδοξία στην Συμφωνία Κορσία πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε στο ETS. Χαίρομαι βεβαίως για το ότι ο ΙΚΑΟ κατέληξε σε μια συμφωνία όταν εγώ και πολλοί άλλοι και η συγκήτρια είχαμε επισκεφτεί τον Νικάο πέρσι υπήρχε μία αίσθηση επιτυχίας όταν καταλήξαμε σε συμφωνία αλλά υπάρχουν τεράστια θέματα όχι μόνο για την φιλοδοξία αλλά και για την εφαρμογή και για το κατά πόσο μπορεί να ε, επιβληθεί σε αντίθεση με το ETS, ε η Κορσία δεν προωθεί τις μειώσεις ε, των εκπομπών, αλλά πρόκειται για μια φιλοδοξία με στόχο ανάπτυξη ουδέτερη ως προς άνθρακα σε σχέση με τα επίπεδα του 2020. Οπότε για οτιδήποτε είναι κάτω από το επίπεδο του 2020 δεν θα γίνει τίποτα. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να αγορά... έχουν τη δυνατότητα οι αεροπορικές εταιρείε να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών και εκεί πέρα θα θέλαμε να εστιάσουμε. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως γιατί ε, πρέπει να υπάρχει η αντιστάθμιση, τα δικαιώματα εκπομπών, αλλά ε, τα αεροσκάφη δυστυχώ σε αντίθεση με άλλα μέσα μεταφορών δεν μπορούν να μειώσουν πολύ τις εκπομπές. Βεβαίως η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, αλλά Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ε, αεροπορία, οι κινητήρες jet ε, δεν έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ από όταν εισήχθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Οπότε πρέπει να δεχτούμε ότι μεγάλο τμήμα θα είναι η αντιστάθμιση των εκπομπών. Το πρόβλημα βεβαίως είναι η ποιότητα αυτής της αντιστάθμισης και το πώς ε, μπορούν να μετρηθεί σωστά. Ο ΙΚΑΟ δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα κανόνες ε, για να ορίσει κριτήρια και όπως επεσήμανε ο εισηγητής η διαδικασία ε, κατάρτισης των κανόνων ε, δεν είναι ούτε δημόσια ούτε έχει διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει στις συζητήσεις. Βεβαίως μπορούμε να λύσουμε διδάγματα από άλλους κλάδους που είχαν τον έλεγχο, την αυτορύθμιση ε, και εκεί ο κάθε κλάδος και βεβαίως στην Επιτροπή εμείς και με το τι έγινε στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι σαφές ότι όταν δεν υπάρχουν ε, επαρκείς ε, έλεγχοι και έχει μια εξουσιοδότηση εν λευκό ο κλάδος οι αποφάσεις δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Βεβαίως θα πρέπει ο κλάδος να εκπροσωπείται και να έχει λόγο τι μπορεί να κάνει ε, από πλευράς ε, μείωσης εκπομπών, αλλά σαφώς η διαδικασία του ΕΚΑ δεν είναι ε, παρκώς διαφανής για να υπάρχει μια εκπροσώπηση όλης της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν θα εξετάσουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, αλλά η Γενική Διεύθυνση Κλίματος ήδη έχει εξετάσει τον μηχανισμό του ΟΗΕ περί καθαρής ανάπτυξης και 73% των αντισταθμιστικών μέτρων του μηχανισμού αυτού από το 2013 μέχρι το 2020 είναι επιλέξει ε, απίθανο να έχουν πραγματικές και μετρήσιμες μειώσεις των εκπομπών. Οπότε αν ληφθούν αποφάσεις να ακολουθεί το μοντέλο, να ακολουθεί το μοντέλο του ΟΗΕ, ε, τίθεται ένα ερώτημα για την ποιότητα αυτών των αντισταθμιστικών μέτρων. Η αεροπορία περιλαμβάνεται λοιπόν σε αυτούς τους στόχους και παραδείγματο χάρη αν η Κορσία αντικαταστήσει ε, το σύστημα της, ε, το ETS εντός της Ένωσης σημαίνει ότι θα είχαμε χαμηλότερους στόχους εκπομπών και αυτό σημαίνει περισσότερο βάρος για άλλους κλάδους. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ πέρα πως στο ψήφισμά μας για τη Συμφωνία των Παρισίων είχαμε πει πως οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας ε, μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν ο μηχανισμός αυτός, ε, δεν λέγονταν τότε κοσέ, είναι φιλόδοξος και αν συνεχίσουν να καλύπτονται οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις από το ETS. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε προφανώς παραβιάζουμε το ίδιο μας ε, το ψήφισμα. Οπότε υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα, αλλά όπως είπα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων. Αλλά οπωσδήποτε θα επικεντρωθούμε σε αυτήν την φιλοδοξία και συγκεκριμένα στην ποιότητα των αντισταθμιστικών μέτρων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερμπράντι τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Τζούλι Γκέρλινγκ ως εισηγήτρια νομίζω πως έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και οπωσδήποτε ε, κάτι που μπορεί να αποτελέσει βάση εργασίας. Σήμερα ξύπνησα και έμαθα ότι ο ε, κλάδος του Χάλιβα είχε αποστείλει μια επιστολή στους υπουργούς και σε εμάς μάλλον λέγοντας ότι βεβαίως είναι υπέρ των κλιματικών πολιτικών αλλά το ETS ε με τη μορφή που συζητείτε τώρα ε, είναι υπερβολικό για την χαλιβουργία. Οπότε, ναι, κλιματικές πολιτικές, αλλά όχι για τη χαλιβουργία. Και το ίδιο ακούμε για το τσιμέντο, για τα λιπάσματα. Με όποια βιομηχανία και αν μιλήσουμε, πάντα το ίδιο ακούμε. Ναι, βεβαίως, αλλά για το δικό μας τον κλάδο είναι διαφορετικά τα πράγματα και είναι αδύνατο να μειώσουμε τις εκπομπές μας. Το ίδιο και με την αεροπορία δηλαδή και ένας πεντάχρονος αντιλαμβάνεται ότι αν πει ο σε αυτό το πράγμα δεν θα πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε ούτε στο Παρίσι ούτε εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Εάν επιμείνουμε στο σενάριο του 1,5 βαθμού των Παρισίων, που πολλοί κόσμος το θέλει, έχουμε τέσσερα χρόνια με τις τωρινά επίπεδα κουμπών και ε, μιλάει για ανάπτυξη ουδέτερη, ουδέτερων εκπομπών η αεροπορία, ούτε καν για μείωση και ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν ε, επιφυλακτικά αισιόδοξο ε, όσον αφορά τη συμφωνία στο Μοντρεάλ και την Κορσία, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ερωτηματικά. Και νομίζω η Τζούλη δικαίως ε, επέλεξε μια επιφυλακτική προσέγγιση απέναντι στον ΙΚΑΟ και την Κορσία. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα που έτρεψαν και από άλλους. Τι συμβαίνει τώρα εντός του ΙΚΑΟ. Πώς πηγαίνει η εφαρμογή του Κορσία. Πώς έχουν τα πράγματα όταν μιλάμε για διεθνείς κανόνες παρακολούθησης και επαλήθευσης. Τι γίνεται με το Μετρό. Τα αντισταθμιστικά μέτρα που αναφέρθηκαν. Απολύτως κρίσιμη σημασία ε, και οι αριθμοί που αναφέρθηκαν ε, βεβαίως ε, από τον συνάδελφο είναι απίστευτοι όσον αφορά το σύστημα του ΟΗΕ. Τα ερωτήματά μου λοιπόν προς την Κομισιόν εντάξει Πρέπει να μας διαφωτίσει λίγο για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο στο επίπεδο του ΙΚΑΟ, αλλά και στο εθνικό επίπεδο μεταξύ των 66 χωρών που έχουν δεσμευτεί να κάνουν πολλά. Τι κάνουν. Συντάσσουν εθνική νομοθεσία για να υλοποιηθεί η κοσία. Και πώς να ερμηνεύσουμε τις επιφυλάξεις κάποιων κυβερνήσεων της Κίνας ειδικότερα για το θέμα της ανάπτυξης χωρίς περαιτέρω εκπομπές. Έχω λοιπόν πολλές ερωτήσεις ακόμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να ακούσουμε βεβαίω τα όσα έχει να πει ο αλλά πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί και να ασκούμε πίεση. Ευχαριστώ κυρία Κιλιώνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω πολύ και την εισηγήτρια για τη δουλειά της, την κυρία Γκέρλινγκ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο καθόλου εύκολο δεν είναι. Οι αεροπορικές ε, μεταφορές αυξάνονται και επομένω οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στον τομέα αυτά αποτελούν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν σχέση και με τα όσα θα γίνουν στο μέλλον στην αγορά των βιοκαυσίμων. Πολλό δε μάλλον που υπάρχει πάντα και μια κοινωνική συνιστόσα. Πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αρκετά και τα κερματισμένος ε, και θα πρέπει να το αναπτύξουμε με συνδυασμένες μεταφορές, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ρωτάμε και μήπως θα έπρεπε να μειώσουμε την ανάγκη για μεταφορές. Ε, εδώ συζητούμε τις αεροπορικές μεταφορές, μας απασχολούν όμως και οι θαλάσσιες μεταφορές ε, και το θέμα είναι πώς θα αντιληφθούν και οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες μεταφορές ε, το μήνυμα του σιδηροδρομικού τομέα. Διότι λέμε όλο ένα και περισσότερο ότι τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται από το σιδηροδρομικό τομέα θα πρέπει να μεταφέρονται με άλλα μεταφορικά μέσα, κάτι το οποίο φυσικά δεν βοηθά στις συνδυασμένες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να πούμε ε, ότι σαφώς και περιμένουμε ε, στο ΔΟΠΑ να προκύψουν κάποιες κοινέ λύσεις, τις οποίες θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλη κλίμακα από κοινού. Αλλά όταν εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, συζητούμε μια πιθανή λύση για τη μείωση των εκπομπών ε, της ναυτιλίας, διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, εάν δεν ε, έχουμε καταφέρει κάποια πρόοδο μέχρι το 2020, δεν ξέρω αν θα αποτελέσουν την καλή λύση. Ε, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε και το ίδιο για τον τομέα της αεροπορίας, να υπάρχουν στόχοι και ε, να δούμε τι θα έχει γίνει μέχρι το 2020 και αν δεν έχουμε καταφέρει τους στόχους να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Ε, πρέπει να γίνουν όλα αυτά διότι ε, ε, πρέπει να υπάρξει μείωση των εκπομπών στον τομέα της αεροπορίας όπως και στην αυτιλία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της COP21 και να ε, σταθούμε στο ύψος των δεσμεύσεων που αναλάβαμε στο παρελθόν Επίσης, ε, θα ήθελα να ε, παρουσιάσω και κάποιες ιδέες, ε, τις οποίες θα μπορούσε ίσως η κυρία Γκέρλιν να αναπτύξει λίγο περισσότερο στην πρότασή της και αφορούν τη βάση συνεργασίας και μέσω της οποίας θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, να γίνονται προτάσεις καινοτομίας, μέτρα δηλαδή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα ωραία και καλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη πολλές φορές ε, δεν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, δεν υπάρχει κατάλληλη ροή πληροφοριών. Όσον αφορά το θέμα της ε, ε, πώληση δικαιωμάτων εκπομπών, πολλά μπορούμε να πούμε στο θέμα αυτό, διότι αν αρχίζουν να συσσωρεύονται χρήματα, για να το πω έτσι, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ναι μεν, αλλά θα έπρεπε τα κονδύλια αυτά να αφιερωθούν στην ε, ενεργειακή απόδοση, ε, στην επένδυση σε καινοτομίε για να αναπτυχθεί η ενεργειακή απόδοση και να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα μοντέλο χαμηλής χρήσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ιδέως σε ένα τομέα όπως είναι οι και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα και στον τομέα της αεροπορίας ε, στην προσπάθεια που κάνουμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ο νέος ευρωπαϊκός ουρανέος. Ναι με ένα απαραίτητο μέτρο αλλά προχωρά πάρα πολύ αργά. Υπάρχει το γεγονός ότι οι εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται όταν πρωτοβουλίες όπως ο ενίος ουρανός θέλανε να μειώσουν τις εκπομπές. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει και τα του οίκου της και να φροντίσει να μειώσει τις εκπομπές στο τομέα της αεροπορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σάικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει μεγάλη ομοφωνία εδώ στην Ομίγυρη και είναι θετικό αυτό, διότι πιστεύω ότι μια κοινή θέση στο Κοινοβούλιο είναι απαραίτητη. Θα μπορούσα να προσθέσω ίσως και ένα-δυο σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Καταρχά να απευθύνω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι συμπεριφερόμαστε όλοι, λες και το Κορσία είναι μια παγκόσμια συμφωνία και όλοι έχουν συμφωνήσει, όταν ξέρουμε στην πραγματικότητα ότι πρόκειται για κάποιες μεγάλες χώρες που έχουν απλώς ε, ε, ε, εκφράσει τις θέσεις τους. Ε, για ανάπτυξη μετά το 2020. Χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, η Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό για αυτές τις χώρες. Θα ήταν λογικό να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το αξιολογεί το θέμα αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε τι να περιμένουμε από ένα μέσο σαν το Κορσία. Εάν υπάρχει μεν το Κορσία, αλλά οι μεγάλες χώρες δεν συμφωνούν καν ε, επί των στόχων, τότε είναι απλώς ένα εργαλείο το οποίο όμως δεν καταφέρνει να επιτύχει ούτε καν τους λιγότερο φιλόδοξους στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και την άποψη της Επιτροπής πριν ε, αρχίσουμε να ε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας ευρωπαϊκής λύσης. Κατά τα λοιπά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γκέρλινγκ, διότι Έλαβα υπόψη τη στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη εγκρίνει στην έκθεση Duncan ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λογικά αυτό κάνει. Βεβαίως εμείς ως πράσινοι θα είχαμε να, θέλαμε να είχαμε πάει έτσι περαιτέρω, να υπάρχει πλήρης δυνατότητα δημοπρασίας για τις εσωτερικές πτήσει. Δεν υπάρχει το φαινόμενο του carbon leakage των εταιριών που φεύγουν και ε, πηγαίνουν αλλού. Ε, μπορούμε να εργαστούμε μέχρι το 2020 μεν, αλλά ξέρουμε ότι μετά το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει και ίδια κάποια μέτρα, που σημαίνει να εφαρμόσουν το κορσία εντό του συστήματο εμπορία εκπομπών. Και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειε και για μα. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγο να έχουμε μια καταληκτική προθεσμία, να σταματήσει το ρολόι και μετά να δούμε ότι και πάλι ο ΔΟΠΑ δεν μα δίνει αυτά που θέλουμε και θα πρέπει να δουλέψουμε μόνοι μα και να αποφύγουμε αυτέ τι επαναλήψει. Αντί να τα κάνουμε, καλό θα ήταν να λάβουμε κάποια μέτρα σε αυτή την αναθεώρηση. Τελευταία παρατήρηση για τις εκπομπές οι οποίε είναι εκτός δοξίδιου του άνθρακα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία καταδεικνύονται από την επιστήμη και χαίρομαι που αναφέρεται στο θέμα αυτό και η συγγήτρια και πάλι, αλλά είμαι ενοχλημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούσαμε τον αντίκτυπο της αεροπορίας ε, από τις εκπομπές εκτός του διοξιδίου του άνθρακα πριν από 7 χρόνια. Στις διαπραγματεύσεις του 2008 το αφαιρέσαμε και μας υποσχέθηκαν ότι θα υποβάλλετε εκθέσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και υπάρχει επιβεβαίωση ότι ο αντίκτυπος της αεροπορίας, αν λάβετε υπόψη και τις μη ε, ε, εκπομπές εκτός διοξιδίου του άνθρακα, είναι διπλάσιος. Ένα αεροπλήνο λοιπόν ε, ε, έχει κι άλλους επιβλαβές εκπομπές και πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη. Τα ξέρετε αυτά, αλλά δεν προτείνετε τίποτα. Επομένως, πότε θα κάνετε κάτι γι' αυτό και χαίρομαι που θα μπορέσουμε τουλάχιστον να το διορθώσουμε με ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα, ώστε να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τις εκπομπές του τομέα της αεροπορίας και όχι μόνο τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο μας είχατε υποσχεστεί το 2008. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης και την εισηγήτρια για το σχέδιο εξαισής Προφανώς και είμαι υπέρ τη ε, φιλοδοξία να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, πολλό δε μάλλον από τον τομέα των αερομεταφερών. Συμφωνώ με τη διαπίστωση των άλλων για τις εκπομπές του οξυδίου του αζότου, ε, των θιούχων αλλά και πολλών άλλων αερούμενων σωματιδίων. Η ομάδα μας ε, είναι αντίθετη στην συμπερίληψη της αεροπορίας στον τομέα, στο σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών, διότι αυτό θα επηρεάσει τις αρμοδιότητες της οργάνωσης της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Εμείς ε, δεν είμαστε κατά ενός μηχανισμού ε, παγκόσμιου της αγοράς, αλλά δεν θα το αποφασίσει μονομερός αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή η αεροπορία είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό τομέα ε, και ορισμένε φορέ οι αεροπορικέ μα εταιρείε είναι θύματα αθέμη του ανταγωνισμού από τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας το ΔΟΠΑ που ε, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χωρών. Κατά συνέπεια λοιπόν διαφωνώ και με τη διάθεση να υπάρχουν ε, ε, δημοπρασίες 50% ε, των εκπομπών για να μειώσουμε το ποσοστό των εκπομπών που δίνονται στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το Euronef και επίσης και την υποχρέωση να δημοσιεύονται αναλυτικά οι ποσοστώσεις όσον αφορά τη δημοπρασία των εκπομπών, των δικαιωμάτων εκπομπών, τα κράτη θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Από νομική σκοπιά, επίση, δεν θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί μέσω πράξεων κατοξουσιοδότηση να καθορίζει τους τρόπους ε, της δημοπρασίας. Ε, Λαμβάνουμε υπόψη μας τα όσα ε, προτείνει ο ΔΟΠΑ και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ότι κάποια από τα πράγματα αυτά αφορούν τη λειτουργία και το χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για μία αρχή η οποία εξαρτάται από τα Ηνωμένα Έθνη, επομένως είναι εξίσου νομιοποιημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και αυτό ολοκληρώνει τον κατάλογο με τους σκιώδεις συγκητές. Θα θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Κυρία Φώστερ, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ελέγξουμε λίγο την πραγματική κατάσταση για το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών ε, στην εμπορία και το πώς δεσμεύει αυτό τις ε, τρίτες χώρες και γι' αυτό πρέπει να βρούμε ένα παγκόσμιο σύστημα Συμφωνώ ότι σε αυτό το οποίο συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε το ρολόι και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι πολύ περιγραφικές κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά αυτό θα πρέπει να κάνουμε να προσφέρουμε την ευκαιρία στη ΔΟΠΑ να συνεχίσει με το έργο της. Τους δώσαμε χρόνια να επανέλθουν με ένα σχέδιο αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι θα λειτουργήσει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι υπάρχουν, υπάρχουν 191 χώρες ε, στην ΔΟΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, εκεί ως μπλοκ και εκτό του παιχνιδιού ε, από πολλές απόψει, Αλλά υπάρχουν άλλε 165 χώρε που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν δεν τι λάβουμε υπόψη και δεν βρούμε κάποια άκρη, τότε δεν θα έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα και έτσι δεν θα είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών. Είναι κάτι που δεν το πετύχαμε τελευταία 12 χρόνια και γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και γι' αυτό πήγαμε στη ΔΟΠΑ για να δούμε αν γίνεται να μας δώσει κάποιες ιδέες για να προχωρήσουμε. Όσον αφορά κάποια άλλα σημεία, είναι πολύ καλό να συζητάμε για τα πρωτόκολλα μη δημοσιοποίηση. Αν κάποιο προσπαθούσε να το κάνει, αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Η ΔΟΠΑ είναι όπως την γνωρίζουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν καλό διάλογο. Υποστήριζω την πρόταση της ε, Επιτροπής πλήρως και υποστηρίζω και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί κατάφερε να πετύχει πάρα πολλά μέχρι στιγμή στο να εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ επάξια Επίσης χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το πώς θέλουμε να δούμε αυτά τα έσοδα. Είναι πολύ αμφίβολο, ασαφές, να, ε, να πιστεύουμε ότι όταν έχουμε έσοδα από τα κράτη-μέλη, έσοδα από τις ευρωπαϊκές εταιρείε, ότι τα πετάμε σε ένα ε, καζάνι που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Όλα τα έσοδα θα πρέπει να ε, ε, χρησιμοποιηθούν για έρευνα ε, στον κλάδο για να προσχωρήσουμε στο μέλλον. Και τέλος, τι θέλω να πω. Δεν έχει νόημα να ελπίζουμε ότι θα πετύχει αυτό το σύστημα δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο σύστημα που θα λειτουργήσει στο Ενωμένο Βασίλειο, που δεν θα είμαστε εδώ μερικά από κάποια χρόνια. Θα είμαστε τρίτη χώρα. Θα ήθελα να πω όμω στα κράτη-μέλη που θα μείνουν ε, ότι πρέπει να είναι προσεκτικά και να προσέχουν τι εύχονται, γιατί έχουμε την καλύτερη ευκαιρία να βρούμε μια συμπεφωνημένη θέση και με την ε, Κίνα και με τη ΣΥΠΑ και όλες τις υπόλοιπες τρίτες χώρες. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω. Ο λόγος που πήγαμε στη ΔΟΠΑ ήταν επειδή κάποιοι σωμάτες όπως το ΕΛΚΑ, το ECR, στην Επιτροπή Μεταφορών θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και φυσικά αναγνωρίσαμε το έργο του κυρίου Λίζε, αλλά στην πολιτική συμφωνούμε να διαφωνούμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε πρακτικοί. Ας ε, συνεχιστεί το θέμα αυτό στο Μοντρεάλ και ελπίζω να βρούμε κάποια ε, συμπέρασματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και ο λόγος στην Επιτροπή έχουμε μαζί μας την κυρία Γκράφ. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Γκέρλινγκ για το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε να ενσωματώσετε όλα τα στοιχεία του ETS σε αυτήν την έκθεση. Εν ώψη της έκθεσης Duncan για την αναθεώρηση του συστήματος ε, δικαιωμάτων εμπορής εκπομπών, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή προτείνει την ε, υιοθέτηση στη ΔΟΠΑ του ψηφίσματος για, την, ε, για το Κορσία. Παρά το ότι είμαστε κάτω από τις αρχικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, μια πολύ θετική εξέλιξη για να θίξουμε και το θέμα των αεροπορικών μεταφορών. μετά την έγκριση τη Συμφωνία του Παρισιού και εν ώψη φυσικά της, αυ... Ε, της αύξησης των ακουμπών στην αεροπορία. Αλλά όπως γνωρίζουμε και πολλοί ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι η έγκριση του ψηφίσματος ήταν ένα πρώτο βήμα και ότι τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να συμπληρωθεί από πολλά στοιχεία που θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την αχαιρότητα του προγράμματος. Γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στην ΔΟΠΑ και αυτό θα καθορίσει την αποδοτικότητα και την ακαιρεότητα του προγράμματος. Κάνουμε λόγο για MRV, για την επιλεξιμότητα μονάδων, για μητρώα, για διπλή μέτρηση και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η διαφάνεια θα είναι βασικό στοιχείο, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην ε, διαχείριση και λειτουργία του προγράμματος και όλα τα στοιχεία αυτά που ανέφερα γι' αυτό. Σας, ε, θα μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στο Μοντρεάλ για να επανέλθουμε στο θέμα του τι συμβαίνει στο Μοντρεάλ, το γεγονό είναι ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει ε, συνεχίζουν και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σύντομα θα μεταφορθούν σε πιο πολιτικό επίπεδο στην ομάδα, στο steering group. Έχουν γίνει κάποιοι πρόοδοι σε διάφορα στοιχεία, σημαντικά στοιχεία, αλλά και άλλα πολλά στοιχεία που είναι σημαντικά για μας είναι ανοιχτά, παραμένουν ανοιχτά και ενδεχομένως ε, θα μας μιλήσουν και πρόβλημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό ως Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της ποιότητας και της ε, ποιότητας ε, των συνθεστικών μέτρων και την ποιότητα των επιλέξιμων μονάδων. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ξεκάθαρη για τις τοποθετήσεις που έχουν ε, οι εταίροι μας σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως είπα ήδη έχουν γίνει συζητήσεις των ε, πυρογνωμών, Κάποιοι δεν ε, μίλησαν, σιώπησαν, όπως η Κίνα παραδείγματος χάρη. και για την ουδετερότητα άνθρακα ως το 2020 και την αρμοδιότητα που έχει η ΔΟΠΑ να εγκρίνει την επιλεξιμότητα κάποιων μονάδων. Κάποιοι άλλοι όπως η Βραζιλία αμφισβητούν ε, κάποια στάνταρ που θέτει η ΔΟΠΑ αλλά πιέζουν, πιέζουν σε άλλα, όπως είναι τα καύσιμα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω για να δούμε πώς αυτές οι χώρες θα τα αντιμετωπίσουν αυτά στην εθνική του νομοθεσία. Ίσως θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η πρώτη δικασία προτού προχωρήσουν σε αυτό και τότε ε, σε εκείνο το διάστημα θα γνωρίζουμε καλύτερα τι θα κάνουν αυτές οι χώρες και αν θα ε, τηρήσουν τις δεσμεύσεις ε, που ανέλαβαν στο Μοντρεάλ. Δύο πτυχέ λοιπόν, ο δικός χάρτης και η εφαρμογή σε ε, ε χώρο επίπεδο. Προφανώς είδατε ότι η πρόταση της έχει λάβει πλήρως υπόψη όλα αυτά και προσπαθεί να διευκολύνει το εναπομείνον έργο στην ΔΟΠΑ, παρατείνοντα ε, το, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογή, άρα έχει την ίδια προσέγγιση και να σταματήσει και πάλι το ρολόγιο. Από την άλλη πλευρά προτείνει να έχει μια αναθεώρηση μόλις θα έχουμε πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα εφαρμοστεί το κορσία. Αυτά είναι τα δύο βήματα. Προτείνουμε λοιπόν, αλλά πρώτα να θίξω και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό και είναι η ανάγκη να εγκρίνουμε γρήγορα μία πρόταση. Γιατί αν δεν ε, εγκριθεί εγκαίρος, τότε θα επιστρέψουμε και πάλι στο πλήρες πεδίο εφαρμογής στην τρέχουσα διαδικασία στην ΔΟΠΑ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη ε, έγκριση μαζί με εσάς και με το Συμβούλιο ώστε να είμαστε εμπρόθεσμοι. Το δεύτερο είναι ότι η τρέχουσα παρέκκληση, παράταση, από την αναθεώρηση θα δώσει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνει τις ε, διεθνείς διαδικασίες και έτσι μόλις θα γνωρίζουμε για τα αποτελέσματα θα προετοιμάσουμε την αναθεώρηση και σε σχέση με την Ίντρα. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, σε βάθος ε, όλα αυτά τα στοιχεία και να δούμε δυνατότητες ε, ε, συμπεριλάβουμε και την ανάγκη να είμαστε συνεπείς ως προς ε, τους στόχους μας και ε, τους στόχους για μείωση εκπομπών που έχει συμφωνηθεί σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνω λοιπόν να αποφύγουμε μια αυτόματη και γρήγορη επιστροφή στο πλήρε πεδίο εφαρμογή. Δεν θα έχουμε τα ε, επιθυμητά αποτελέσματα σε διεθνέ επίπεδο και θα μας ε, φέρει σε πολύ δύσκολη θέση κάτι τέτοιο. Ας έχουμε υπόψη ότι πάντα μπορούμε να αλλάξουμε κάποια χαρακτηριστικά όταν προετοιμάζουμε την αναθεώρηση. Πέρα από αυτά ε, μας αρέσουν οι τροπολογίες που πλαισιώνουν καλύτερα την αναθεώρηση και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθούμε σε κάποιους προβληματισμούς για το μέλλον και παράλληλα Πιστεύουμε ότι το σύστημα εκπομπών μετά το 2021 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην επόμενη αναθεώρηση, εξολόγηση και αυτό που περιμένουμε είναι να υπάρξει μια προβλησιμότητα για τους ε, χειριστές και να υπάρξει και μια συνεπία στο 2030 και τους στόχους που έχουν τεθεί για τότε. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μαζί σας και για όλα τα στοιχεία της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέρλινγκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, τέτοια ώρα που είναι δεν θα τα αναφέρω όλα. Έχω σημειώσει τα όσα ακούστηκαν. Είναι πολύ καλή η ομάδα των σχεδόν εισηγητών. Προβλέπω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τα αποτελέσματα του Κορσία. Εγώ δεν βλέπω εναλλακτική άλλη πέρα από αυτό το οποίο σας είπα εγώ. Υπάρχει μόνο μια εναλλακτική, δηλαδή να επανέλθουμε στο προηγούμενο του ETS. Και χαίρομαι που κανείς δεν προτείνει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα αυτό πρέπει να το δύο ο ως μια κίνηση εξαιρετικά θετική και ελπίζω στο πνεύμα αυτό να δεχτούν ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες πληροφορίες που θα θέλαμε, λίγο περισσότερη διαφάνεια και φιλοδοξία. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς εδώ πάμε προς την σωστή κατεύθυνση. Αναμένω βεβαίω και τις ε, τροπολογίες των συνάδελφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για τροπολογίες είναι 7 Ιουνίου στις 11 και ψηφίζουμε στις 11 Ιουλίου. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.